ανακοίνωση από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα μου ανακοίνωσαν ότι διορίζεται στην Επιτροπή Προϋπολογισμών ο κ. Γκονζάρες Πόνς αντικαθιστώντας τον κ. Ιτουργκάης. Υπάρχουν